Υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες ε, σε σχέση με την ασφάλεια και χρειαζόμαστε μία νέα προσέγγιση ούτω ώστε να ομαδοποιήσουμε τους διάσπαρτους νομοθετικούς πόρους, αν θέλετε, που έχουμε και να έχουμε ένα διατομεακό διάλογο ε, για όλες τις ε, θαλάσσιες δραστηριότητες και να χρησιμοποιήσουμε το διάλογο χρησιμοποιώντας πιο συγκεκριμένα υψηλότατα πρότυπα Χρειαζόμαστε μια βιομηχανία που να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια ούτω ώστε να γνωρίζουν όλοι τι γίνεται. Χρειαζόμαστε φεδρικά σχέδια επίσης ε, για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ε, και ε, τρόπους αντιμετώπισης των ατυχημάτων χρησιμοποιώντας δημόσιους πόρους ή οργανισμούς όπως ο ΕΜΣΑ αλλά και άλλοι ούτω ώστε αν χρειαστεί και ταχύτατα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε από μια θαλάσσια περιοχή μια άλλη θαλάσσια περιοχή σε περίπτωση ατυχήματος. Έχει εργαστεί πάντως και η βιομηχανία για να υπάρχει ο διαθέσιμος ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Επίσης, σας είπα ότι αυτό που ενδιαφέρει όλους τους φορείς είναι να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές και τα ατυχήματα και η διάθεση των πόρων ε, να αναλαμβάνεται από την ε, εκάστοτε αρμόδια αρχή ε, και να καθαρίσουμε το ταχύτερο δυνατόν οποιαδήποτε πέτρελαιο κοιλίδα. Ο Ριπένον πληρώνει. Νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί αυτήν την αρχή, αλλά πρέπει να δούμε και το θέμα της αστικής ευθύνης και να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να υπάρχει μία ισορροπία ανεξαρτήτως κλίμακος του φορέα εκμετάλλευσης δηλαδή. Επίσης επανειλημμένα έχουμε συζητήσει το θέμα του ότι ε, Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολλές χώρες που συνορεύουν με την Ένωση και εύκολα μπορούν να επηρεαστούν ε, από πετρελαιοκυλίδες και το αντίστροφο. Αυτό ισχύει για τη Μεσάεως για τη Βαλτική, τη Βόρεια Θάλασσα κτλ. Οπότε δεν ε, ε, αρκεί η δέσμευση μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε, στις διασυνοριακές, ε, στις μεθοριακές μάλλον περιοχές. Όσον αφορά τις τροπολογίες θα γίνουν και κάποιες άλλες συζητήσεις για την αδειοδότηση και για τους μηχανισμούς στην Ένωση. Ένα από τα σχόλια που κάναμε είναι πως θα πρέπει να εφαρμοστεί ό,τι νομοθεσία και να συμφωνήσουμε και η Κομισιόν θα πρέπει να προσέχει τα της επιβολής. Οπότε συμβαίνουν ε, πολλά και διάφορα. Κάποια μπορεί, απλά να συμπληρώνουν ε, τρύπες στο παζλ της νομοθεσίας και βέβαια υπάρχει και το θέμα της διεθνούς συνεργασίας. Προσωπικά, έχοντας παρακολουθήσει κάποιες από τις συνεδριάσεις στην ε, Κομισιόν με ρυθμιστικές αρχές ε, σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές. Βλέπουμε πως υπάρχει πολύ καλή δουλειά σε διαφορετικά ζητήματα που επηρεάζουν τη βιομηχανία και όπως σας είπα υπάρχουν απλά όλες οι ρυθμιστικές αρχές που συναντιόνται για να υπάρξει μια συνεργασία βεβαίως και η ίδια η Κεντρική Ρυθμιστική Αρχή, όπως έχει πει, δεν έχει την δυνατότητα να πάει σε κάποια μεμονωμένη εγκατάσταση πετρελαίου ή αερίου. Λοιπόν, ε, αναμένω τη συνεργασία με τους κοιότε ηγητές και είμαι σίγουρη πω θα έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χόλ έχει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν στην αρχή της ε, παρουσίασης. Είμαι ευγνώμων στην εισηγήτρια για την καλή συνεργασία που είχαμε και υπάρχουν ε, πολλοί τομείς τους οποίους νομίζω πως έχουμε καταλήξει σε μια συνένεση όσον αφορά το τι είναι σημαντικό από πλευράς ασφαλείας, την σημασία της επαλήθευσης από τρίτα μέρη, την έγκαιρη ενημέρωση και τη διαφάνεια όσον αφορά τυχόν περιστατικά για να μοιράζονται οι πληροφορίες άμεσα. Τρία σημεία εγώ θα αναφέρω ε, τα οποία νομίζω ότι είναι κάπως ε, σημαντικά. Πρώτα απ' όλα για το θέμα της ε, εποπτείας. Και ε, νομίζω πως μιλάμε για το ίδιο πράγμα με την εισηγήτρια. Σαφώς υπάρχει μία ανάγκη να πάμε πέρα από ένα εθελοντικό σύστημα συνεργασίας γιατί σε τελική ανάλυση αν μια εταιρεία δεν τηρεί τις ε, προδιαγραφές αυτό έχει φοβερές και εκτεταμένες συνέπειες, αλλά αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει πρόβλημα δυναμικότητας και θα μπορούσαμε να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα εάν προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε ε, ένα επίπεδο στο ευρωπαϊκό επίπεδο πέρα από τα ήδη υπάρχοντα. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποια υποχρεωτική εφαρμογή γιατί τίποτα λιγότερο δεν θα διασφαλίσει την εφαρμογή των απαιτήσεων, αλλά εμένα με ενδιαφέρει το μοντέλο του Μπέρικ που έχουμε στις επικοινωνίες όπου συναντώνται οι ρυθμιστικές αρχές και γίνονται έτσι ε, ένας ε, επιπλέον ρυθμιστικός φορέας. Οπότε το θέμα είναι ένα συντονισμός και όχι ένα επιπλέον επίπεδο που θα περιπλέξει τα πράγματα. Όσον αφορά την αρκτική αντιλαμβάνομαι όσους ε, εκφράζουν ανησυχίες για το πόσο ευάλωτη είναι η Αρκτική, αλλά η πραγματικότητα είναι πως υπάρχουν ήδη ε, εγκαταστάσεις εκεί πέρα, οπότε πρέπει να τονίσουμε την ιδιαιτερότητα της εξόριξης ε, στην Αρκτική και να τονίσουμε πως ε, θα έχουμε ειδικέ απαιτήσει που θα διασφαλίζουν πως η εξόριξη στην Αρκτική ε, γίνονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ειδικά το πόσο ευάλωτες είναι αυτές οι περιοχές πρέπει να ληφθεί υπόψη οπότε Πρέπει να πάμε πάρα πέρα, να σκεφτούμε ευρύτερα από ό,τι θα κάναμε οπουδήποτε αλλού. Και τέλος, θεωρώ πως πρέπει να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί όσον αφορά τη λειτουργία ευρωπαϊκών εταιριών στα στα παγκόσμια ύδατα. Ε, πρέπει να δούμε το τι γίνεται σε, άλλες, σε άλλους κλάδους, σε άλλες βιομηχανίες όσον αφορά πολυεθνικές εταιρείε και γίνονται προσπάθειες με το να υπάρχει αναφορά από χώρα σε χώρα για να υπάρχει διαφάνεια. Νομίζω πως ε, έχουμε μια υποχρέωση ως νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουμε πως οι εταιρείε με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ε, εφαρμόζουν επικίνδυνες και τσαπατσούλικες ε, τακτικές σε άλλα μέρη του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ η κυρία Καρβάλιο. Thank you very much, President. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγγήτρια τη Βίκη Φόρντ. Ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία μας. συμφωνήσαμε για θεμελιώδη ζητήματα και υποβάλαμε και μια σειρά τροπολογιών που συνυπέγραψαν ο εισηγητής και οι εισηγητές. Έχουμε δηλαδή επιτελέσει την, ε, το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς μας για τις συμβαστικές τροπολογίες. Υπήρξε πάρα πολύ καλός συντονισμός ανάμεσα σε όλους τους εισηγητές. Είχαμε ανησυχίες σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της έκθεσης και λήφθηκαν υπόψη όλε, όλες οι παρατηρήσεις μας σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες που όπως σας είπα συνυπέγραψαν οι σκιώδεις και η συγγήτρια. Ε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό αναφέρουμε τώρα, ενώ το αρχικό σχέδιο απέδει ένα σημαντικότερο ρόλο στα κράτη-μέλη, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εάν συμβεί κάποιο ατύχημα στην Βόρεια Αφρική, παραδείγματο χάρη, ε, θα επηρεάσει και τις χώρες της Νοτιού Μεσογείου. Οπότε χρειαζόμαστε συνεργασία για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχα και ένα άλλο ε, σχετικό σχόλιο σε σχέση με την ΕΜΣΑ, δηλαδή τον Οργανισμό για την ε, Ασφάλεια στις Θάλασσες. οφείλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο της για την πρόληψη των ατυχημάτων. Ήδη λειτουργεί ένας ε, μηχανισμός, δηλαδή εντοπίζουν ε, την πετρελοκυλίδα λίδα ε, στα πλαίσια του μηχανισμού πρόληψης των ατυχημάτων που οφείλονται σε σκάφη ε, δηλαδή ήδη στην αρχή ε, της καταστροφής του ατυχήματος από μια πλατφόρμα εξόριξη εντοπίζουν πολύ γρήγορα την ε, πετρελαιοκυλίδα και άρα υπάρχει ταχεία ανταπόκριση διότι λειτουργεί ένας μηχανισμός βάσης το οποίο διάφορα σκάφη περιπολούν και καλύπτουν ε, όλα τα χωρικά ύδατα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα οποιοδήποτε ατύχημα σχετίζεται με πλατφόρμα εξόρυξης καλύπτεται. Τρίτον, χρειαζόμαστε σαφέστερο ορισμό περί δημοσίας ευθύνης. Συμφωνώ πολύ με τη Βίκη. Η βιομηχανία δηλαδή θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο της για την αστική ευθύνη. Αυτό το στοιχείο υπήρχε στην αρχική έκθεση. Τώρα τονίζουμε το ρόλο του δημοσίου τομέα για θέματα ασφάλειας συντονισμού ε, ως προς την ανταπόκριση περίπτωση ατυχήματος και προσδιορίζουμε πακριβέστερα τα καθήκοντα που θα επομιστούν οι δημόσιες αρχές. Ε, εν μια άλλη παρατήρηση τώρα που βάλαμε στο δεύτερο σχέδιο. Το πρώτο σχέδιο βασιζόταν στη μεγάλο βαθμό σε εμπειρίες που, εμπειρίες που είχαμε από την Βόρεια Θάλασσα για την μεταφορά τεχνογνωσίας από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τη Βόρεια Θάλασσα και τη μεταφορά λοιπόν της τεχνογνωσίας προς άλλες ε, περιοχές. Και αυτό το στοιχείο πλέον συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο της έκθεσης. Τελευταία παρατήρηση. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείε να ε, λειτουργούν βάσει των ε, ιδίων προτύπων ασφαλείας ε, ανεξαρτήτως χώρου δραστηριότητας. Μπορεί να είναι οπουδήποτε στην Ιφίλιο. Αυτό το στοιχείο δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο και ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια, την Βίκη Φόρντ γιατί δέχτηκε και ενσωμάτωσε τις θέσεις μας καθώς και τις θέσεις των υπολείπων σχεδόν εισηγητών ήταν πολύ ευχάριστη η συνεργασία με τη Βίκη Φόρτ και με τους υπόλοιπους σκιώδες εισηγητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ενά. Ευχαρι... Κύριε Ενά. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Χθες ε, συζητούσαμε για την οδηγία σε Βέζο 3 και από τους... Ε, έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, συμμετείχαν οι βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες και σημειώσαμε πρόοδο. Τώρα βρεθήκαμε σε άλλο πλανήτη σήμερα. Ε, οι κανονιστικές ρυθμίσεις ε, αδυνατούν να αναβαθμίζονται και δεν μπορούν να ακολουθήσουν την, τις ραγδαίες εξελίξεις στη βιομηχανία. Υποθέτω ότι δεν θα συζητήσουμε την τροπολογία της ΕΒΕΖΟ 3 γιατί είναι άχρηστη. Ούτως ή άλλως τα κανονιστικά συστήματα αδυνατούν να εξελιχθούν. Ε, πρέπει να εγγυηθεί η ασφάλεια και των μισθωτών και του περιβάλλοντος και των πολιτών και θα κάνω λοιπόν μια πολύ απλή πρόταση. Η πετρελαιοβιομηχανία θα πρέπει να υπαχθεί στους κανόνες Εβέζο 3. Αυτό θα ρυθμίσει πάρα πολλές δυσκολίες και όταν μας λένε ότι ναι μεν αλλά μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα μα το αντίθετο. Καμία πετρελαϊκή εταιρεία δεν ναι, το έχει κάνει ποτέ αυτό ε, πέρσι στη Γαλλία 10 δις ευρώ κέρδη είχαν, άρα δεν νομίζω δεν έχουν λεφτά για να πληρώσουν ε, τους ελέγχους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σκίνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω Θέλω να ευχαριστήσω του δύο συγητέ που με βοήθησαν πάρα πολύ να βρω τη σωστή ισορροπία σε αυτή την έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω και, τις, και την εισηγήτρια για την ε, πολύ καλή δουλειά που έκανε και που είχε δίκον ούς για τις συμβολές των σχεδόν εισηγητών. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία είπαμε νομίζω τα έχει λάβει υπόψη, αυτό είναι θαυμάσιο και μας δίνει πολύ καλές ελπίδες για το μέλλον πρέπει να κατανοήσουμε ότι όταν γίνεται υποθαλάσσια εξόριξη έχουμε πολλές χώρες από μας έχουν μεγάλη εμπειρία για τα θέματα αυτά και επομένω δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε ιδιαίτερη εμπειρία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζονται πρόσθετες στρώσεις γραφειοκρατίας για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως οι διαρροές και τα αρνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον που μπορούν να προκύψουν από ε, δυσκολίες, από αστοχίες σε εγκαταστάσεις σε, σε εξόριξη σε βαθαία ύδατα. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα για τη συνεργασία των κρατών μελών, αλλά ως εκεί μονάχα. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία θα ήθελα να συμπεριληφθούν στην έκθεση και δεν έχουν συμπεριληφθεί. Ίσως υπάρχουν κάποιε φιλοσοφικέ διαφορέ στα θέματα αυτά. Εγώ θα ήθελα να υπάρχουν ανεξάρτητε εκθέσει ε, ασφαλεία. και επίση πιστεύω ότι η οδηγία για τα μηχανήματα θα μπορούσε να καλύπτει και τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε πλατφόρμες εξόρυξης και αν ληφθούν υπόψη όλα αυτά που περιλαμβάνονται στην οδηγία του ΣΕΒΕΖΟ και στην οδηγία για τα μηχανήματα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και αυτά έχουν κάποιες ε, επιπτώσεις για τις εξορίξεις στο βυθό της θάλασσας. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ισχύουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ώστε να υπάρχει η εγγύηση ασφαλείας όλων των εμπλεκομένων. Χαίρομαι λοιπόν που η συγγήτρια έχει δείξει μεγάλη σοφροσύνη και έχει λάβει υπόψη όλων και από τη δική μας πλευρά είμαστε έτοιμοι να την υποστηρίξουμε και στη συνέχεια τη διαδικασίας. Σας ευχαριστώ. Μερσή λέει ο Πρόεδρος. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν κ. Σάνεκ έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους τους εμπλεκομένους στη διαδικασία αυτή. Κατανοώ ότι υπάρχουν πολλά επιτεύγματα τα οποία υπάρχει η αίσθηση ότι έχουν επιτευχθεί πολλά στην έκθεση αυτή και επίσης υπάρχει και το θέμα της συνένεσης η οποία έχει επιτευχθεί και εμείς ήμασταν πάντα στη διάθεση όλων για στοιχεία πληροφόρησης και ελπίζω ότι σας έχουμε δώσει επαρκή στοιχεία πληροφόρησης για όλα τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια συγκλίνουσα άποψη που εστιάζει σε μερικά βασικά σημεία που έχουν να κάνουν με την ε, ασφάλεια των εξορίξεων σε βαθαία ύδατα. Ο στόχος μας είναι να υπάρχει μια νέα όθηση που θα δοθεί και, στην, και στον κλάδο ε, των εξορίξεων και στους ε, επόπτες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι συνεχίζεται η η προσπάθειά μας και με την έκθεση αντικτύπου και επίσης όλα αυτά θα αντανακλώνται στις πρωτοβουλίες που θα φέρει η Κομισιόν ενώπιον στους επόμενους μήνες και από τις ε, απόψεις που ακούστηκαν σήμερα διαπιστώνω ότι υπάρχει κάποια ανησυχία σε σχέση με την ε, προσθήκη πρόσθετων στρωμάτων γραφειοκρατίας για τα θέματα αυτά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η πρόθεσή μας να επιβάλλουμε επιπλέον διαδικασίες, να δημιουργήσουμε ένα περιττό άχθος για τον εξορρυκτικό τομέα. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν αποδείξιμη προστιθέμενη αξία, εμείς δεν έχουμε πρόθεση να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οι αναλύσεις τις οποίες έχουμε προβεί Βέβαια, έχουμε δείξει ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύτερα από ότι σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο μεμονωμένων εταιριών. Θα εστιάσουμε την προσοχή μα εκεί και μόνο Συμφωνούμε επίσης ότι θα έπρεπε να καταστεί δυνατό για τον Ευρωπαίο νομοθέτη να δημιουργήσει ένα κλίμα, μια κατάσταση όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν σε όλο τον πλανήτη θα είναι υποχρεωμένες να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα και τήρηση των κανονισμών από τις εταιρείες αυτές. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα θέματα της ε, εξοεδαφικότητος αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πολύ έδαφο για θελοντικούς κώδικες συμπεριφοράς. Και τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι και πάλι αναφέρθηκε η έκφραση της εποπτείας των εποπτών, του ελέγχου των ελεγκτών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε τώρα όλη αυτή την αντιμετώπιση και να την αντιμετωπίσουμε εκτός πλαισίου. Υπάρχουν πολλές δράσεις οι οποίες προτείνονται στην έκθεση αυτή και μας δίνουν τρόπους να έχουμε μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν αποτελεσματικά ότι η λειτουργία των ελεγκτικών αρχών θα υπόκειται σε δημόσια επιτήρηση και έλεγχο των ε, μέσων που χρησιμοποιούνται ώστε να βρίσκονται στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο, ώστε επομένως να υπάρχει δυνατότητα οι ελεγκτές να είναι υπόλογοι και ελέγξιμοι προς το καλό των Ευρωπαίων πολιτών. Και φυσικά παραμένουμε στην ε, διάθεση της εισηγήτριας και των σκιωδών ώστε να σας δώσουμε και πρόσθετες πληροφορίες εφόσον αυτό το ζητήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φόρτ για να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι γιατί δεν ήταν εδώ όλοι οι σκιώδες. Στην αρχή, αρχή είπα σας ευχαριστώ εσάς, ε, τους συμβουλούς σας, ε, τους βοηθούς σας, όλοι όσοι συνέβαλαν σε, αυτή τη δουλειά. Τέλο υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν πίσω μας, δίπλα μας, μας βοηθούν. Όλους τους ευχαριστώ. Τώρα, σε σχέση με αυτά που μας είπε ο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, φυσικά θα χρειάζεται καλό συντονισμό ούτως ώστε να έχουμε επαγγελματική αριστεία από πλευράς όλων ε, των ρυθμιστικών αρχών. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες ε, από τις παρατηρήσεις. Για την Αρκτική, συμφωνώ ότι όλοι όσοι κάνουν εξόριξη με τρόπο που ενδέχεται να πλήξει το περιβάλλον πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσουν τις βέλτιστες ε, πρακτικές ε, και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Αρκτική αλλά και στη Μεσόγειο. Οπότε πιστεύω πως ε, θα πρέπει να μεριμνήσουμε για να ισχύουν υψηλότατες προδιαγραφές ασφαλείας και το αναφέρω αυτό διότι σε κάποια θαλάσσια ε, περιβα... υπάρχουν ευαίσθητα θαλάσσια περιβάλλοντα σε διάφορες περιοχές, όχι μόνο στην Αρκτική. Ε, ε καταλαβαίνω αυτά που λέτε για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τα ίδια όμως θα πρέπει να ισχύουν και για τις μη ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ε, διότι ούτως ή άλλως όταν εκπονούμε την νομοθεσία λαμβάνουμε υπόψη τις εξελίξεις ανά τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε από την εμπειρία των άλλων αν ε, δραστηριοποιούνται ε, κάποιοι χωρίς να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας ε, θα είναι ευπρόσδεκτοι στο βαθμό που θα εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες. Ευχαριστώ κυρία Καρβάλιο για τις παρατηρήσεις σας. Έχετε επισκεφτεί την ΕΜΣΑ και μας προσφέρετε την εμπειρία που αποκομίσατε και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. τώρα για, τις, για τις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου συμφωνώ ε, και μιλήσαμε για την περίπτωση της Νορβηγίας ε, και σε μία από τις τροπολογίες, συμβαστικές τροπολογίες το αναφέρουμε. Δηλαδή, βασική προτεραιότητα στην εξόριξη είναι η ασφάλεια και το προσωπικό πρέπει να το ξέρει και δεν πρόκειται μόνο για νορβηγικό μοντέλο και σε άλλες πλατφόρμες εξόρυξης ε, ακολουθούν το ίδιο σύστημα. Αυτή είναι η διαφορά. Θα ήθελα επίσης να θυμόμαστε ότι όταν μιλάμε για εξόριξη υψηλής πίεσης. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ε, σε βαθιά νερά στην ανοιχτή θάλασσα. Μπορεί να έχουμε ατύχημα ε, λόγω της υψηλής πίεσης ε, που θα είναι επικίνδυνο και για το θαλάσσιο περιβάλλον ε, και για τις ανθρώπινες ζωές σε βαθύ ύδατα. Οπότε όταν μιλάτε για υπεράκτια ασφάλεια να έχετε κατά νου ότι δεν είναι ασφαλή όλα τα βαθύ ύδατα ούτε επικίνδυνη η ανοιχτή θάλασσα εν και θέλω να το επιθυμίσουμε σε όλους τους συναδέλφους γιατί είναι εύκολα, εύκολα πέφτει κανείς αυτή την παγίδα. Στην Νορβηγία, παραδείγματο χάρη, ο τελευταίος κίνδυνος ε, που απετράπη ήταν σε βαθύ ύδατα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Κλείσαμε λοιπόν με την ημέρα διάταξη για σήμερα. 16 Ιουνίου θα ε, γίνει ψηφοφορία. Πάμε στο σημείο 13. Έχει να κάνει με, τα, με τις δημόσιες, δημόσιες συμβάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνω το λόγο στον κύριο Σιμάνσκι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάνει μια γνωμοδότηση για την έκθεση ε, Ρούλε η οποία είναι η συγγήτρια επί της ουσίας στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Έχω ανακανοισμένες παρατηρήσεις για τα θέματα των δημοσίων συμβάσεων από την οπτική γωνία της βιομηχανίας και των βιομηχανικών κλάδων. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια στο δίκαιο και να μην υπάρχουν συνεχείς αλλαγές όπως αντιμετωπίζουμε τώρα τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των ε, κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη διοικητική εργασία και τη διαχείριση αυτών των διασημοσίων διαχωνισμών, κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα για τις μικρομεσαίες ιδιω επιχειρήσεις, διότι οι, μικρές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χάνουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στους δημόσιους διαγωνισμούς λόγω των προβλημάτων αυτών διοικητικού χαρακτήρα. Γι' αυτό η εστίαση στην δική μου γνωμοδότηση εστιάζει στο πρόβλημα αυτό και αναφέρεται σε μια έρευνα που έγινε στις Ηνωμένε Πολιτείες σε σχέση με τους δημόσιους διαγωνισμούς και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σωστή κατεύθυνση, είναι ένα υπόδειγμα το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Το δίκαιο για τους δημόσιους διαγωνισμούς θα πρέπει να μας ε, βοηθήσει να επιτύχουμε άλλους σημαντικούς στόχους όπως είναι η καινοτομία, η αποδοτικότητα στη χρήση της ενέργειας, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κτλ. Και επομένως το σύνολο αυτών των στόχων στον τομέα των δημοσίων διαγωνισμών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν με αυτή οι στόχη χωρίς να βλάψουμε την ανταγωνιστικότητα, δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικό αποκλειστικά τα κριτήρια και δεν θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος την δυνατότητα να διαλέγουμε πάντα αυτόν ο οποίος προσφέρει την πιο ελκυστική τιμή. Είναι σημαντική λοιπόν η τιμή η οποία προσφέρεται στους διαγωνισμούς και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Ένα άλλο δεύτερο σημαντικό κριτήριο είναι και η αναγκαιότητα να υπάρχει μια λεπτομερής ε, έκθεση αξιολόγησης κάθε φορά πρόμιας αποφάσεως θα πρέπει να σκεφτόμαστε και για άλλους στόχους που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, όπως είπα προηγουμένως, με την καινοτομία. Και μόνο όταν λάβουμε υπόψη αυτούς τους ε, κανόνες θα μπορούσαμε να έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση. Αυτά είναι λοιπόν τα βασικά στοιχεία της γνωμοδότησης τα οποία εγώ ήθελα να σας παρουσιάσω. Και η ελπίδα μου είναι ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και την υποστήριξη όλων των συναδέλφων για την ε, γνωμοδότηση που πρέπει να δώσουμε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε η κυρία Χολ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας στις δημόσιες προμήθειες που αναφέρεται στην εκθεσή σας. Είναι πολύ σημαντικό, έχει τονιστεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Φεβρουάριο στο σχετικό σχέδιο της Κομισιόν πως οι δημόσιες προμήθειες έχουν να παίξουν μεγάλο ρόλο στο να κινητοποιήσουν την αγορά για τέτοια προϊόντα και να συνεισφέρουν στο να έχουμε εξοικονόμηση ενέργεια στην Ένωση. Επίσης σημαντικό είναι να τονίσουμε πως υπάρχει και τεράστια οικονομία γιατί αυτό απασχολεί πάρα πολύ με την οικονομική κρίση οι αρχές έχουν μειωμένους προϋπολογισμούς και σημαντικό είναι να θυμόμαστε πως το να αγοράζουμε τέτοια προϊόντα πρόθεσμα ήδη θα έχει σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Η PricewaterhouseCoopers και η Ecofis έκαναν μία μελέτη κόστους κύκλου ζωής το 2009 που έδειξε πως οι πράσινες δημόσιες προμήθειες θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 20 δισεκατομμύρια ε, τη, στην Ένωση. Και βεβαίως οι πράσινοι είναι λογιστές, δεν είναι καμία πράσινη μικιό. Οπότε καλό θα ήταν να τονίσουμε στη γνωμοδότηση το πόσο σημαντική είναι αυτή η πτυχή όχι μόνο από τη ζωτική σκοπιά εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και λόγω του, της εξοικονόμησης που θα φέρει. Επίσης συμφωνώ με τον κύριο Κρότσμαν που είναι εδώ αυτή τη στιγμή πως πρέπει να φροντίσουμε οι διαδικασίες δημοσίων προμηθειών να είναι σαφείς ώστε να μην εμποδίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλουν προφορές για υπηρεσίες και αγαθά που αγοράζει ο δημόσιος τομέας. Εάν έχουμε κάποια απλοποίηση, νομίζω πως θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία. Παρακάτω, Μπένσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρειάζεται ο εξυγχρονισμός ε, των δημοσίων προμηθειών. Έχουμε πολύπλοκους κανόνες και είναι δυσκίνητη η διαδικασία για τις αρχές και άρα ε, ακριβή για τους φορολογούμενους και βεβαίως υπάρχει και βάρος διοικητικό στις μικρόμεσες επιχειρήσεις. Υπήρχαν πολλές αποφάσεις του ΔΕΚ ε, και άρα υπάρχει μια νομολογία που πρέπει να λάβουμε υπόψη για να είναι σαφείς οι κανόνες. Συνολικά πιστεύω πως ο κύριος Σιμάνς έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο πλαίσιο της γνωμοδότησης. Θα ήθελα όμως η γνωμοδότηση να δώσει περισσότερο βάρος στην απλοποίηση και μείωση του διοικητικού βάρους καθώς επίσης και το να ρίξει βάρος το πώς θα δώσουμε καλύτερη πρόσβαση στην διαδικασία υποβολής προσφορών και συμφωνώ που θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τους κανόνες δημοσίων προμηθειών όχι μόνο ε, όσον αφορά να εξετάζουμε τον μειοδότη αλλά να το δούμε πιο μακροπρόθεσμα και να έχουμε βεβαίως και κατά νου τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας. Αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να μην καταλήξουμε με νέες διοικητικές απαιτήσεις για τις αρχές και ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να γίνουν έτσι πάλι ακριβές οι δημόσιες και να αποθαρρύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης πρέπει να φροντίσουμε να μην εισαχθούν κριτήρια για να ε, μπορούμε να καταλήξουμε έτσι μόνο σε εθνικούς υποψηφίους. Επίσης, όπως ανέφερε και η Φιώνα, χρειαζόμαστε περισσότερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η καλή δουλειά της Κομισιόν με ένα κώδικα βελτίστων πρακτικών για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να λυθεί όταν εξυγχρονίζουμε τους κανόνες δημοσίων προμηθειών. Στο ψήφισμα περί μικρών επιχειρήσεων που υιοθετήσαμε πριν από δύο εβδομάδες είπαμε πως θέλουμε να ενισχύσουμε τον διάλογο μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό που κάνουν τις αγορές του δημοσίου. Πρέπει να γίνει αυτό, να δούμε πώς θα ενισχυθεί αυτός ο διάλογος, χωρίς βεβαίως να μειωθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πλευράς κομισιών. Θέλει κάποιος να μας εξηγήσει κάτι. Όχι. Να δώσω το λόγο πάλι στον κύριο Σιμάνσκι. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αρκετά ευρεία συνένεση στην Επιτροπή μας και συμφωνώ ότι η ενεργειακή απόδοση είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για το νέο δίκαιο και περί κρατικών προμηθειών. Για την γνωμοδότηση τώρα, πρέπει να καταδείξουμε την ανάγκη εξέβρεση ισορροπία ανάμεσα σε αυτή τη διάσταση και άλλε εξίσου κέρυε διαστάσει για τι κρατικέ προμήθειε. Είμαι πεπισμένο ότι μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση για να εκφράσουμε τη βούλησή μα, την πρόθεσή μα να ενσωματώσουμε και αυτή τη διάσταση στη νέα νομοθεσία περί κρατικών προμηθειών. Η σαφήνεια τώρα του δικαίου είναι απαραίτητη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό αναφέρθηκα στο αμερικανικό πρότυπο και στην ανάγκη ε, επίτευξης πολύ μεγαλύτερης σταθερότητας. Γιατί νομίζω ότι το πλέον επιζήμιο στοιχείο για τις ε, μικρές κυρίως επιχειρήσεις αυτό είναι στο ε, ε, δίκαιο, στο εργατικό δίκαιο. Και το μόνο ε, που χρειάστηκε να κάνω είναι να ε, περικόψω την αρχική μου ε, έκθεση αλλά τώρα πια μπορούμε να προσθέσουμε λεπτομέρειες, να αναπτύξουμε το θέμα και θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες βασιζόμενος στις δικές σας και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε συνένεση στην Επιτροπή ganz Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει μια σημαντική ανακοίνωση, 15 Ιουνίου, 12 η ώρα. Προθεσμία για τις τροπολογίες. Κανείς δεν έχει αντίρρηση, οπότε ελήφθη και αυτή η απόφαση. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, γιατί οι ψηφοφορίες προβλέπονται για τις 10. Οπότε σας ανακοινώνω πως μπορείτε να πιείτε ένα καφεδάκι. Αλλά παρακαλώ 10 η ώρα να είστε εδώ. We start with boat, because we have so many boats.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ψηφίζονται αυτό μαζί. Μετά, θα πει ο Πρόεδρος του Ρεσμού Ελεμένου της Ελλήντα, out of courtesy, συνήθως δεν κάνουμε, δεν κανείς. Ωστόσο, όταν πάει στην πληροφορία, εμείς είμαστε εναντίον. Ήταν αυτό που συζητήσαμε χθες. Objection, συνήθως out of courtesy, δεν σήκωνε κανείς χέρι και πάμε κατευθείαν στην πληροφορία. Εντάξει. Και σας, σας τα έχω στο σημείο.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 Yeah. Come. Yeah. Come. Meine Damen und Herren, liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι λέει ο πρόεδρος, κυρίες καθώς και κύριοι, φίλοι, δεν με ακούει κανένας λέει ο πρόεδρος. <laughs> Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, γιατί έχουμε μπόλικες. Και ορισμένες από αυτές τις ψηφοφορίες θα είναι δύσκολες, πολύπλοκες. Όχι μόνο πολλές ψηφοφορίες, αλλά κάπως δύσκολες κατά σημεία. Χρειάζομαι λοιπόν τη βοήθειά σας και την επίοικια και κατανόησή σας. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική πρώτα ψηφοφορία για να ξέρουμε καταρχήν ποιοι είναι παρόντες, ποιοι δεν είναι παρόντες και αν δουλεύει το σύστημα. Ψηφίζουμε για το κατά πόσο στο μέλλον θα ξεκινάμε εγκαίρως. Θα πείτε ναι, όχι ή αποχή παρακαλώ. Ξεκινάμε. 47 ήμασταν, λείπουν ορισμένοι όμως. Αλλά δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, όλα δουλεύουν. Εντάξει, no problems. Κυρία Μαδουρέλ, έχετε πρόβλημα. Δεν πειράζει. Α, πέρασε ψηφοφορίες, δεν προφθαίνετε να ψηφίσετε. Δεν μπορείτε πια να ψηφίσετε. πλούι, δεν μπορείτε να ψηφίσετε άλλο σήμερα το πρωί. Αυτή είναι η κανόνη the new rule. Who missed the first vote, that's all. Λοιπόν, ξεκινάμε με την έκθεση Jordan Σίζελη διαχείριση εξαντλημένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων τροπολογίες 47 και 50 από κοινού 47 και 50 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτονται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. Ποιοι είναι κατά καταρχήν για την 3. Μπορείτε να ξεσηκώσετε χέρια στις αποχές. Γίνεται δεκτή. Τροπολογία 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Θεέ μου, λέει ο πρόεδρος. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Άρχεται, είπα. Δεν δουλεύει. Τώρα, εντάξει. Ξαναψηφίστε, παρακαλώ. Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Πάλι από την αρχή. Μα τι γίνεται εδώ πέρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας από το ΕΛΚ περισσεύει. Ένας πράσινος περισσεύει. Είναι όλα εντάξει τώρα, πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Δεν βλέπετε το αποτέλεσμα. 31-19 ήταν το αποτέλεσμα. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 και 9 μαζί υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος έλεγχος 8 και 9 μαζί άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται 24-27. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές δεκτή 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 152 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 153 υπέρ κατά αποχές Απορρίφθηκε. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 και 154 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές επίσης δεκτό. 1.55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά Μπορώ να το ξανακάνω αυτό. 18 ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 1.59 και η 19 μαζί. Εκπίπτουν 158. Εκπίπτει και αυτή. Ωραία. 160. 160 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Απόχε. Δεκτή. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 130 και 131 καθώς και 17 καθώς και 14 που είναι όλες ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτές 132 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ εκπίπτει, εκπίπτει, εκπίπτει α, συγγνώμη εκπίπτει γιατί είναι κρίθη 132 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1-3-3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 136 και 140 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 137 και 15 ως προστίκες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 138 με χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ συγγνώμη εκπίπτει μόνο το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ εκπίπτει εκπίπτει διότι εκρήθη 20 ναι 11 και εδώ και εδώ εκπίπτει και 141 το ίδιο και 139 επίσης 143 και 21 που είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 144 καθώς και 22 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 145 Καλύπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 εκπίπτει. Κατά συνέπεια 163 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα 20 του, της ηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατόν 68 εκπίπτει. Όχι, 168. Την ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ για την 168. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1,67. Υπέρ. Εκπίπτει. Ωραία, ευχαριστώ. Σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα. 170 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ άρχεται Πέρας. Απερίφθη. Με μικρή διαφορά. 24-26. 21. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ. Έλεγχος για την 21. Ζητείτε. Θέλετε έλεγχο. Α, δεν το κατάλαβα. 21 έλεγχος. Άρχεται. 21. Ψηφίσουμε την 21 ηλεκτρονικά για έλεγχο. Η 21. Και πάλι από την αρχή. 21 κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 21. Αρχίσει η ψηφοφορία. Για βάση, για βάση, να προλάβουν όλοι. 21 του περιβάλλοντος ή του, της εισηγήτριας. Της εισηγήτριας. <laughs> της εισηγήτριας. Πέρασε. Πέρας. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. Αμ. Έτσι δεν πρέπει να αμφιβάλλετε για την, για την κρίση μου, μου φαίνεται, μετά από αυτό. 173. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 177 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ τα αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 καθώς και 22 ένδυ και 25 ε, έμπλ ψηφίζουμε κατά αποχές απορρίπτονται 100 τσεκ βεβαίως μα ήταν σαφές αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία Άρχεται. Ένας από το ΕΛΚ περισσεύει. Ένας από το ΕΛΚ πρέπει να σταματήσει να ψηφίζει, όχι να βγει από ναι, την να μην ψηφίζει απλώς. Ευχαριστώ, πέρας. Απορρίπτονται. Κύριε Βιτικόφερ, δεν έχω πάντα δίκιο, αλλά συνήθως έχω. Συνήθως έχω. 181 και 23. Ένβη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27. Έμπλ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές δεκτή 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 184 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 183 υπέρ κατά δεκτή 28 εκπίπτει ευχαριστώ 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 εκπίπτει 23 και αυτή πέφτει. Πέφτει και η επόμενη, πέφτει και η επόμενη. Εκπίπτουν. Πηγαίνουμε στην 5. Όχι. I think 201, 201 νομίζω είναι η επόμενη. Μια στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία στη γραμματεία. Rapporteurs, okay. 102 choose next one. 174. 174, 174. Because we have 187. a Ah, Ms. Rapporteur is right. 174. 174 είναι η επόμενη. Εντάξει, έχει δίκιο η γραμματεία. 174. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα που πάμε 201 λέει ο πρόεδρος My God, is that complicated? <laughs> Uh, no, 193. 193, okay. 193, λέει ο πρόεδρος. 193 ψήφι υπέρ. Υπέρ, κατά, απόχες, δεκτή. 194 υπέρ, κατά, άποχες δεκτή. 199 εκπίπτει. 200 εκπίπτει. 201 εκπίπτει επίσης. Καταπίπτει και 201. Εκατόν Συγγνώμη, είναι πεπλεγμένα τα πράγματα. 197 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για την 197. Έλεγχος ηλεκτρονικός στην 197 άρχεται. One Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Ε, okay. Now, ein bitte. Ένας από το ΕΛΚ να μην ψηφίζει παρακαλώ. Jetzt, weil es keine, so wenig Kompromisse gibt, deshalb. Alles klar? Ein EPP zu viel, da muss jetzt mal... Περισσεύει κάποιο από το ΕΛΚ. Λοιπόν, αποφασίστε ποιο θα ψηφίσει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Πέρα ψηφοφορία εγκρίνεται. Εκπίπτει 195, 196, 24, 198. 25. 25 Ψήφι υπέρ της 25. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ. 26 υπέρ και πάλι. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 206. Εκπίπτει. 206, όχι, δεν, δεν εκπίπτει. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 207, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 208, υπέρ. Κατά και πάλι 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε έλεγχο στη 208 έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία Δύο πράσινοι πέραν του ορίου. Αυτό αρχίζει να γίνεται εγκληματικού χαρακτήρα εδώ πέρα. Μήπως θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πιτικό εκτός μικροφόνου. 208. Okay now? 208. Εντάξει. Πέρασε. Εγκρίνεται. Μπράβο. Ωραία. 209 εκπίπτει. 30. Απασχόληση υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 210 καθώς και 31, καθώς και 27 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία έλεγχο. Πέρας. Απολύπτονται με ισοψηφία 25-25 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2-12 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 εκπίπτει 2-13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2-14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές απολύπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.15 υπέρ κατά αποχές απολύπτεται. 2.16 καθώς και 33 καθώς και 31 ψήφι υπέρ κατά εποχές απορρίπτονται. Θέλετε έλεγχο βεβαίως. 2, 16, 33 και 31. Πάμε. Άρχεται. Εντάξει. Πέρας. Εγκρίνονται. 34. 34. 34 υπέρ. Όχι, όχι. 34 υπέρ. Και πάλι θέλετε. Μπορούμε να απορρίψουμε την προηγούμενη άμα θέλετε. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.19 καθώς και 32 και 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Κάπως καλύτερα πάντα τα πράγματα. 2, 32 και 35 ηλεκτρονικός ελεγχο τώρα. Πάλι. 219, 32 και 35 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία. Εντάξει, πέρας. Απορρίπτονται. Δύο, είκοσι, τριάντα τρία και τριάντα έξι. Η 216 δεν απερίφθη όμως. η 216. Άρα πρέπει να τις ψηφίσουμε, λέει η γραμματεία. Yeah, a question was 22. I must Yeah, Yeah, that was my credit. 22 and 32. 220. 33 και 36 ψήφοι υπέρ υπέρ κατά έλεγχος έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία άρχεται And the vote is closed. Απορρίπτεται. 2.17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.22 καθώς και 34 ένβη εκπίπτουν. Βεβαίω. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.23 εκπίπτει, 2.24 καθώς και 35 ένβη, καθώς και 38 έμπου, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.25 εκπίπτει, 2.26 σαν προσθήκη υπέρ, κατά, Αποχές δεκτή 27 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. 2.27 έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 2, 28, 36, ένβη, 39, έμπλου είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 2,29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για τη 40 άρχεται άμα πέρας εγκρίνεται 2.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.33 με 37 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 2.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 έμπλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 28 και 27 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 2.35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 2.36 καθώς και 39 ένβη με τμήματα, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα. Χωρίς τη λέξη final υπέρ κατά πάλι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα α θέλετε έλεγχο καλά πρώτο τμήμα ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας εγκρίνεται Συγγνώμη, έκανα λάθος. Άμα δείχνετε τα χέρια σε όλοι δεν θα είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερο τμήμα εκπίπτει. 42 εκπίπτει.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 κατά αποχές εγκρίνεται 40 NV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 εκπίπτει δεν μπορεί κανείς να συνεχίσει έτσι είναι πάρα πολύ πολύπλοκα όλα αυτά 44 κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.39 εκπίπτει πάμε στη 47 της απασχόλησης ναι, οι 240, συγγνώμη, 240 και 46 είναι ταυτόσιμες, ψηφίζουμε. 240 και 46, κατά. Αποχές εγκρίνονται. 47, υπέρ κατά αποχές απορρίβεται 31 ναι είναι τα ε, συμβατή υπέρ έλεγχος 47 έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται σαφές. 31 υπέρ κατά δεχτή 2.42 υπέρ κατά άποχες νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά δεν είμαι σίγουρος 2.41 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Χωρίς τη λέξη existing. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα με τη λέξη existing. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης συγκρίνεται. Η 41 εκπίπτει, 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε. έχονται αυτές που μου αρέσουν, συμβαστικές. Συμβαστική τρία Υπέρ. Κατά. Αποχές. τρία αλφα συμβαστική. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τι όμορφα που είναι. Φεύγουμε. Έφυγε όλη η σελίδα. 33 και 250 από κοινού. Ψήφι υπέρ κατά <clears throat> αποχές εγκρίνονται 2.49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 2.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.52 όχι όχι όχι όχι λέει η γραμματεία έχει εγκριθεί η 33. 2-53, 2-54, 2-55. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 34 ψηφίσουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκριθεί. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 256 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 έλεγχος για τη 256 άρχεται έτσι έτσι <laughs> Περάσε. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται με ισοψηφία. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 ΕΝΒ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 NV υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 έμπλη υπέρ κατά αποχές δεκτή 259 εκπίπτει Δύο εξήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δύο εξήντα ένα υπέρ. Όχι, για εκπίπτει, συγγνώμη. 2,62 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 2,63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2,64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος. Για τη 264, παρακαλώ. <clears throat> Άρχεται. Εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. 37 και 36 με χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, όπως έχει τροποποιηθεί προφορικά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Με προσθετή φράση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το 36 είναι το ίδιο με το 37. Τα ψηφίσαμε μαζί. Εντάξει. 265 εκπίπτει, 266 εκπίπτει, 67, 66, 67. Πάμε σε 268. Υπέρ. Κατά αποχέ υπέρ της 268 λέει και πάλι ο πρόεδρος κατά αποχές απορρίπτεται 269 εκπίπτει 38 την ψηφίσουμε τι 38 είπε, είπε 38 πρόεδρος συγγνώμη 38 ψηφίζουμε 38 Την 38 την ψηφίσουμε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2,70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 εκπίπτει. 2,71 και 48 που είναι ταυτόσιμες ψηφίζουμε ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται εκπίπτει 41 41 υπέρ κατά εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 έμπλε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.74 υπέρ Κυρία Φαν Μπρέμτ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να προτείνω μια προφορική τροπολογία λέει η τροπολογία στο δεύτερο μέρος ε, υψηλή προτεραιότητα θα δοθεί σε παλαιά ραδιενεργά απόβλητα επειδή υπάρχει δυνατότητα παρεξήγησης αντί να πούμε ε, παλαιά να πούμε τα παλαιότερα Keiner, alle einverstanden, all agree. Εντάξει, συμφωνείτε όλοι. 2.74 με την προφορική τροποποίηση που έχει κάνει η Καθλίν Φαν Ψήφι υπέρ. Κατά. ...2.74 με την προφορική τροποποίηση, σας λέω και πάλι ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. εκπίπτει 42 ψήφι υπέρ κατά ψηφίζετε ή όχι μήπως μπορείτε να ψηφίσετε ποιοι είναι υπέρ ε, ευχαριστώ μερσή κατά αποχές εγκρίνεται 278 εκπίπτει εκπίπτει 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 44 υπέρ κατά δεκτή 281 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.85 υπέρ κατά δύο ογδόντα πέντε υπέρ κατά από εγκρίνεται 45 καθώς και 286 που είναι ταυτόσιμες ψήφοι υπέρ κατά από εγκρίνονται 287 εκπίπτει 50 288 288 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 289 υπέρ. Εκπίπτει. 290-291. Ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 292 σε δύο τμήματα και με προφορική τροποποίηση. Ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματο. Κατά αποχέ δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Εκπίπτει. Α, κρίμα. 2,93 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 7 έμπλη υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά 54 υπέρ πάλι από την αρχή 54 υπέρ Excuse me. Once again, number 7 in check. 7 ample check. Vote is open. 7 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. All voted. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρασε. Adopted. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 εκπίπτει, 58 εκπίπτει, 59 έχει αποσύρθει, 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 <clears throat> υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ένα ένβη υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 έμπλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ένα της ηγητρίας υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα καλύπτεται Εκπλήτω το πρώτο τμήμα δεύτερο τμήμα Ψηφιπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 εκπίπτει, 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 70 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 74 εκπίπτει. 73 επίσης. 71 και 72 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Πάλι από την αρχή. 71 και 72 υπέρ Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Έλεγχος. Εντάξει. Αν δεν δείχνουν τα χέρια δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Μόνο αυτούς που σηκώνουν τα χέρια τους μπορώ να μετρήσω. Δεν μπορώ να μαντέψω τι κάνουν οι υπόλοιποι. Πέρας. Εγκρίνονται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο περιβάλλον. Έχει εκπέσει. 76. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος βεβαίως έρχεται ο στο πρώτο τμήμα πρώτο τμήμα της 76 πέρας απορρίπτεται δεύτερο τμήμα της 76 εκπίπτει 77 εκπίπτει, 78 επίσης, 78 ε, <clears throat> την ψηφίσουμε παρόλα αυτά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 79 καθώς και 3 NV ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ε, έλεγχος, έλεγχος. Λοιπόν, άμα είναι έτσι, να κάνουμε συνέχεια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αλλιώ σηκώνετε τα χέρια σα. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία 79 και 3. Πέρασε. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Τι είπατε. Εκτός μικροφώνου σχόλια. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 85 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. 85 έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 85, την είπαμε τώρα, ναι. Και 84 εκπίπτει. 87. Δεύτερο τμήμα. 84, το δεύτερο τμήμα μόνο να ψηφίζουμε. Εντάξει. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 87. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 MV υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά άποχες δεκτή 90 υπέρ κατά αποχές απόλυτοτε. Γίνεται 91 εκπίπτει. Συμβαστική 1 υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ υπέρ κατά αποχές απόλυτοτε. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εκατό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, οι 12 και 6 είναι ταυτόσιμες, ψηφίζουμε κατά, έχουν εκπέσει όμως. Έχουν εκπέσει. Πέσανε. 103 υπέρ. Κατά. Κατά παρακαλώ σηκώστε πάλι τα χέρια σας. Αποχές απορρίπτεται. 7 <clears throat> ένδυ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 106 έχει... Ε, η 8 υπέρ. Κατά. Η 106 είχε αποσυρθεί. Οχτώ ένβη υπέρ πάλι. Κατά. Απόχειας δεκτή. Ε, συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ο Αλάχ λέει ο πρόεδρος. 11. 11 ένβη. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τσεχ έλεγχος έντεκ, ένδυ. Έντεκα επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 109 υπέρ συγγνώμη εκπίπτει εκπίπτει ναι 112 πάμε 110 υπέρ κατά 110 υπέρ κατά έλεγχος 110 άρχεται η ψηφοφορία Πέρασε. απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά Συγγνώμη πρέπει να κάνουμε έλεγχο 115 Άρχεται Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία ελέγχου στην 115. Πέρας. Εγκρίνεται. 116 εκπίπτει. 6. Εισηγήτρια. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117. Εκπίπτει. εκπίπτει 12, 118, εκπίπτει 7, Επτά της εισηγήτριας υπέρ κατά έλεγχος στην επτά. άρχεται άρχεται πέρασε απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ α εκπίπτει 122 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 122 Απόλυτα. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 NV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 ως υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ Σαν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και η τελειωτική κυρία Σίζελη <clears throat> ε, μην σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που είναι μακρύτατος ο κατάλογος της ψηφοφορίας, αλλά διαπιστώνεται το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουμε για αυτό το θέμα και παραμένει λίγα αναμφιλεγόμενο. Ε, προσπαθήσαμε πραγματικά πάρα πολύ με τους σκιώδεις εισηγητές για να καταλήξουμε συμβαστικέ τροπολογίε. Δυστυχώ μόνο σε τρει καταλήξαμε. Μετά λοιπόν από τη μακρά ψηφοφορία αντιλαμβάνομαι ότι όλοι κέρδισαν κάτι αλλά, όλοι έχασαν και κάτι. πολλέ τεχνικέ λεπτομέρειε κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία και εξού και οι απορρίψει των τροπολογιών. Ζητώ να υποστηρίξετε την οδηγία διότι χρειαζόμαστε ισχυρότατη πλειοψηφία ενώ ενώπιον του Συμβουλίου. Ε, ε, δεν, έπρεπε, δεν έπρεπε να το έχω επιτρέψει. Συγγνώμη, όχι, ήταν λάθος, ήταν λάθος μου, δεν θα το επαναλάβω όμως, όχι δεν θα ακούσουμε, άλλως θα ψηφίσουμε σοβαρά. Όχι, συγγνώμη, ήταν λάθος μου, ζητώ συγγνώμη, ήταν λάθος μου, ε, κύριε Πρόεδρε κάνει και κακή δουλειά και την επενείται και δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα. Ε, δεν χρειάζονται προσβολές λέει ο Πρόεδρος. Ήρεμο κλίμα δεν είναι ανάγκη να συγχύζεστε. Μία ώρα ψηφίζουμε, επιτέλους πρέπει να τελειώσουμε. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. And the vote is closed. Πέρας. Και εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος. Ναι, 33 υπέρ, 6 κατά 12 αποχές, μα το βλέπετε. Δεν, ναι, δεν έκανα λάθος. Και τώρα ψηφίζουμε επί του νομοθετικού ψηφίσματος. Συμφωνείτε. Άρχεται η ψηφοφορία. Νομοθετικό ψήφισμα. Πέρας. Και... Τα αποτελέσματα εγκρίνεται και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πέρας. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. δεν, δεν θα ξαναγίνει το ίδιο πράγμα. Όχι πάρα πολύ συχνά παρακαλώ αυτό το πράγμα. Και σας ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες και όσο πιο ήρεμοι είστε τόσο πιο γρήγορα θα πάνε τα πράγματα. a δεν γίνονται, δεν γίνονται όλα μαζί. Πόσους να ακούω κι εγώ. Εάν υπάρχει κάτι, πείτε μου όταν φτάσουμε. Αν θέλει να πει κάτι ο εισηγητής, έχει τώρα την ευκαιρία. Κύριε Χατζημαρκάκη, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι πέρα από την... Ε, σε αντίθεση με την άλλη έκθεση, έχουμε πολλές συμβαστικές τροπολογίες, θα κυλήσουν γρήγορα τα πράγματα και υπάρχει άλλη μια συμβαστική τροπολογία που δεν υπάρχει στον κατάλογο, στη σελίδα υπαριθμών 5. Η υπαριθμών 14α η συμβιβαστική. Κάποιες τροπολογίες καταπίπτουν εκεί. Δεν είναι σημειωμένοι Ήθελα να σας το πω, η γραμματεία θα σας ειδοποιήσει όταν φτάσουμε εκεί. Λυπούμε. Δεν αναφέρεται εδώ, αλλά θα γίνει η δουλειά μας πιο εύκολη. Να δούμε, λέει ο πρόεδρος. Θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παριθμών 10 υπέρ. Κατά. Α, ήδη άρχισα τα λάθη. Λίγη ησυχία παρακαλώ, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είμαι σε φόρμα. 137 υπέρ. Κατά. Μα δεν είπατε. Πώς ζητάτε πάλι, δεν είπα καν το αποτέλεσμα. Πιο γρήγορη από τον ήχο. Δηλαδή, ξεπερνάτε και τον εαυτό σας πια. Ο Κλόντ πυροβολεί πιο γρήγορα από τη σκιά του. Λοιπόν, να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ein check eines Boat is open. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι λιγότεροι εδώ πέρα, ναι. Άρα, πέρας. Εγκρίνεται. δέκατη συμκοϊπέρ κατά αποχές δεκτή 141 υπέρ κατά αποχές δεκτή ποιος, τι επαλήθευση συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 149 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 161 δεν ψηφίζεται. Σωστά, σωστά. 12 της ΕΚΟΝ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 της κατά καταπίπτει. 165 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 166 υπέρ Ορίστε. 165. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. 165 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ιδέα του κυρίου Τούρμες. Πέρας της ψηφοφορίας. Και κύριος Ρόιλ έχει σαφή πλειοψηφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τα χρειάζομαι αυτά πρωί-πρωί, έτσι, θαυμάσια. Να το επαναλάβουμε. 166 πέρ. Κατά. Ε, κάπως λίγη. Αποχές δεκτή. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 13 έκον υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. 168 υπέρ. Ε, επαληθεύσουμε, συγχωρείτε. Τέρας. Και απορρίπτεται. 169. Τι Α, Έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 13 ε, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά απορρίπτεται νομίζω συμβαστική 14 κατά αποχές δεκτή 189 υπέρ κατά αποχές δεκτή 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά απορρίπτεται λοιπόν, να επαληθεύσουμε την 20 Closed. Πέρας, δεκτή. 191 πίπτη 19 υπέρ. Κατά. Να ξαναδώ ποιοι είναι υπέρ. Ωραία, ευχαριστώ, δεκτή. Συμβαστική 14α. Την έχετε μπροστά σας, δεν την διαβάζω. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή καταπίπτουν όλα αυτά μέχρι την 192 ψηφίζουμε την 192 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τώρα τι γίνεται με την επόμενη να επαληθεύσουμε την 192 ε χρόνος υπάρχει 192 επαληθεύουμε Και πέρας. Ε, λίγο πιο γρήγορα. Πέρας δεκτή. Ε, σωστές 196 μέχρι 199 ε, έχουν τακτοποιηθεί όλα αυτά καταπίπτει 216 ταυτόσιμος φέρ κατά Έκανα λάθο. Η 199 δεν κόλλαγε. Α. 199 υπέρ. Τα αποχέ δεκτή. 216 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ. Κατά. αποχέ δεκτή. 201 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. «22 και 202 υπέρ». Λάθος. Α, καταπίπτουν. Α, κάποιος μου είχε πει ταυτόσημες. Α, καταπίπτουν. 203. 203 υπέρ κατά αποχές δεκτή 204 υπέρ κατά αποχές δεκτή 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ απορρίπτεται 15 της εκών υπέρ κατά αποχές δεκτή 206 περ κατά αποχές δεκτή 207 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή Δύο 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 229 υπέρ κατά Δύο ξανά υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές Να επαληθεύσουμε. 2.30 υπέρ. Ε, 2.30 με συγχωρείτε. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο τριάντα ένα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 232 κατά πίπτη, 233 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 234 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 235 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 236 καταπίπτει. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 έκον υπέρ κατά αποχές δεκτή. 242 υπέρ κατά να το επαναλάβω 242 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Ε, συγγνώμη, εγκρίνεται. 243 και 19 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 27 και 244 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.45 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.52 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η επόμενη καταπίπτη. 23 τσίμκο υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 μκο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτή. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 265 υπέρ. Κατά. Να παληθεύσουμε. 265. πέρας δεκτή 26 της υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 20α υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές 31 υπέρ κατά απορρίπτεται 32 υπέρ κατά δεκτή 20 συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 της έκον υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.73 υπέρ κατά αποχές δεκτή 43, 34 υπέρ κατά αποχές 35 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε 35 Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά έχει δεκτή. 2,85 υπέρ. 2,78 μισχόρτη υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2,79 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2,80 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2,81 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.84 πίπτη 2.85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές 38 υπέρ κατά αποχές 2,87 υπέρ κατά αποχές συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές 2,92 υπέρ κατά αποχές συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 24β υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 3.11 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 312 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 26 καταπίπτει, 313 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 3, 14 και 27 υπέρ κατά αποχές δεκτές 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3, 16 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε 3.16 Πέρας Απορρίπτεται 3.17 υπέρ Κατά Να επαληθεύσουμε 3.17 Πέρας. Δεκτή. 3.18 υπέρ. Κατά. Να δω ποιοι είναι υπέρ. Ναι, ναι, δεκτή, δεκτή. 3.19 υπέρ. Κατά. έχεις δεκτή. Σαφής, σαφής λουσία. Να επαληθεύσουμε την 319. Αν θέλετε. Πέρας. Ναι, δεκτή. 320 υπέρ. 321 υπέρ κατά αποχές να δω ποιοι είναι υπέρ 321 κατά αποχές δεκτή 322 καταπίπτει 323 υπέρ κατά αποχές δεκτή 324 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβατική 25 υπέρ κατά δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 334 υπέρ κατά αποχές δεκτή μα υπέρ ψηφίσανε καλώς 3.34 να την επαληθεύσουμε. Closed. Πέρας. Απόρριπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτή. 32 έμκο υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά ξανά υπέρ παρακαλώ 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.51 καταπίπτει ή 28 συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1 υπέρ έκον κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 62 και 63 υπέρ κατά αποχές Ναι, δεκτή θα έλεγα κι εγώ. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 66. Ψηφίζουμε ή καταπίπτει. 69. 69. 69 υπέρ, κατά Νομίζω δεκτή. Ορίστε. Να επαληθεύσουμε. Νομίζω ότι ήταν δεκτή. Να Πέρασμα. Πέρας, στην επαλήθευση ψηφίζουν λιγότεροι πάντα. Δεκτή. Στην πέμπτη ψηφοφορία είμαστε μόνοι. 2 υπαριθμών 2 καταπίπτει 4 καταπίπτει 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Συγγνώμη, άρχεται. Εβδομήντα δύο. Πέρας. Και απορρίπτεται. Εβδομήντα τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές δικτύ. Τρία καταπίπτει. Εβδομήντα τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81, 82, 83 υπέρ. 83. τρία υπέρ. Κατά. Υπαριθμόν 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκτή. 85 υπέρ. Κατά Βαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 92 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 93, 94 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 95 υπέρ. Κατά πιπτή. 96 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 ψήφου υπέρ κατά αποχές δεκτή 97 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4β υπέρ κατά αποχές δεκτή 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή 102 υπέρ Κατά. εποχές απορρίφθεται Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. εποχές δεκτή. 4 υπέρ. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 117 υπέρ κατά αποχές να υπαλληθεύσουμε την 117 εγώ νομίζω ότι έχει υπερψηφιστεί πέρας απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή 123 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 και 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή καταπίπτουν 125 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε Πέρας. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 134 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 135 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 135 να επαληθεύσουμε την 135 Πέρας. Απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία, άρχη ψηφοφορία. rejected. Και απορρίπτεται. irgendwas ε, νεράκι παρακαλώ. Λοιπόν. Είναι η μέρα του μαρτυρίου, λέω. Τι, τι, τώρα. Όλα αυτά.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 on or not? No? No? Yes? Okay. Τώρα. 119 ε, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 121. Τι, τι τρέχει με το μικρόφωνο. 121 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ να επαληθεύσουμε την 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 129 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 130 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 130 να την επαληθεύσουμε. Άρχεται. Την 130, 130 μου ζητήσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. Καλό είναι όσοι είναι εδώ να ψηφίζουν. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά καλό. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 18 της Ρέγγι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 142 υπέρ κατά αποχές δεκτή 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 151 υπέρ κατά αποχές 152 υπέρ κατά αποχές 153 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε 153 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Rejected. απορρίπτεται 154 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.29. Καταπίπτει. 2.29 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 5 της Ρέγγι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 305 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 155 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 169 υπέρ κατά ξανά 169 υπέρ κατά Αποχές. Να την δούμε. Την 169 επαλήθευση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 9 της Ρέγκη υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 172 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε 172 άρχεται πέρας απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές δεκτή 174 υπέρ κατά αποχές δεκτή 175 υπέρ κατά αποχές δεκτή 176 υπέρ κατά αποχές δεκτή 177 υπέρ κατά αποχές δεκτή 150 υπέρ κατά αποχές δεκτή 478 υπέρ. Καταπίπτει. Με συγχωρείτε. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 203 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές 216 πέρ κατά να επαληθεύσουμε την 216 216 Closed. Πέρασε. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2.33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.35 υπέρ κατά αποχές δεκτή ρέγγι 4 υπέρ α καταπίπτει καταπίπτει καταπίπτει ρέγγι 6 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε Άρχεται η ψηφοφορία. And... Πέρας και δεκτή. Εγκρίνεται λοιπόν. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 2.52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.53 υπέρ κατά αποχές δεκτή Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και δεκτή. 2.54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 20 υπέρ αποχές δεκτή επίσης 2.71 ξέχασα κάτι 2.71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.73 υπέρ κατά 2.73 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορριφθείτε, αλλά να επαληθεύσουμε. Να είμαστε σίγουροι. 2,73. Πέρας και απορρίπτεται. 2,76 πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 21. Υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 22 υπέρ κατά Εποχές δεκτή συμβαστική 23 υπέρ κατά Εποχές δεκτή 24 υπέρ κατά Εποχές δεκτή 25 υπέρ Κατά. αποχές δεκτή 3-12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 313 υπέρ κατά αποχές δεκτή 314 πίπτη 315 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 322 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.42 υπέρ κατά δικτή. δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.53 υπέρ κατά αποχές δεκτή 354 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 362 υπέρ κατά αποχές δεκτή 363 υπέρ κατά Να επαληθεύσουμε. 363. Άρχεται η ψηφοφορία. Eine Karte zu wenig, Pech gehabt. Λείπει μια κάρτα, ατυχήσατε. Τέλος πάντων, ναι. Και θέλετε υπέρ ή κατά. Κατά να ψηφίσετε, δεν έχει σημασία. Κατά. 364 υπέρ κατά αποχές δεκτή 365 υπέρ κατά αποχές δεκτή 366 υπέρ κατά αποχές δεκτή 367 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε 367 Συνένα. one. Closed, Απορρίπτεται. Συμβαστική 37. Υπέρ. Κατά. Ναι. Αποχές. Δεκτή. Wonderful pages. Τι θαυμάσια σελίδες. Μπράβο. 375 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 376 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4.28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4.29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 300 καταπίπτει ρέγγι 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 464 υπέρ κατά αποχές δεκτή 465 υπέρ κατά αποχές δεκτή καταπίπτει 467 465 να επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας και εγκρίνεται. 467 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 468 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τέσσερα, 68 να την επαληθεύσουμε, είναι ευκολότερο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 472. 72 υπέρ. Κατά. αποχέ Δεκτή. 473 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. 474 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. 474. Άρχη τη σοφορία. Και... Πέρας. Απορρίπτεται. 4,75 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 4,76 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4,77 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4,79 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Πέρας. Όχι απορρίπτεται. 4,80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορριφτεται. 4,81 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4,82 υπέρ. Και 83 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. Closed. Wieso? Du musst doch dafür stimmen, das ist doch deine eigene Scheiße. Πέρας. Ναι. 484. Ορίστε. Το αποτέλεσμα ήταν 24 κατά και 18 υπέρ. 24 με σχόλιο υπέρ και 18 κατά. Μα, μα τι, τι ψήφισε ο ίδιος. Κοιτάξτε. Ε, τόση ώρα που ψηφίζουμε έκανα, έκανα και λάθος και καταψήφισα τη δική μου τροπολογία. Αφού σας χαροποιεί, ορίστε. Ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως θα είχε απορριφθεί. 4.84 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 4.85 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε 4.85 Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 26 περ. Κατά. Εποχές δεκτή. 496 περ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δύο κομμάτια στην 47 Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ Κατά. Ε, Κάπω χειρότερα. Νομίζω απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Ρέγγι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4,98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4,99 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 504 υπέρ κατά αποχές check να επαληθεύσουμε ε, προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά... Closed. Πέρας. Ναι, απορρίπτεται. 504 υπέρ κατά μα το όχι 505 υπέρ κατά εποχές 207 507 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές 517 υπέρ κατά Α, δεν υπήρχε καν. 515 515 5-15 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5-16 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές Ρέγγι 7 υπέρ κατά αποχές δεκτεί, Ρέγγι 24 υπέρ κατά δεκτεί, δεκτή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέγγι 16 καταπίπτει 5-30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 Θα ψηφίσουμε τώρα για την 16 ε, της περιφερειακής, Ρέγγι 16. Κατά. Α, ε, απορρίπτεται. 5.30. Κατά. Απορρίπτεται. 5.31. Κατά. Απορρίπτεται. 532 υπέρ κατά εγκρίνεται 533 καθώς και 534 ταυτόσιμες υπέρ κατά εγκρίνονται 535 κατά εγκρίνονται. Ρέγγι 25. Όχι. Εκπίπτει. 536. Υπέρ. Κατά. Κατά. 536 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 30 κατά εγκρίνεται 544 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα κατά εγκρίνεται δεύτερο τμήμα κατά δεν εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα 545 εκπίπτει συμβαστική 31 ψήφι Εγκρίνεται 548. Κατά. χανε, Από την... Απορρίπτεται 555. Υπέρ. Κατά. Πέντε, πέντε, πέντε υπέρ. Κατά. 556 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 557 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 558 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 559 κατά εγκρίνεται. Η ρέγγι 15 εκπίπτει. Συμβιβαστική 32. Κατά. Εγκρίνεται. Ρέγγι 10. Κατά. Εγκρίνεται. 560 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Κατά. Απορρίπτεται. 570. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 571 και κατά εγκρίνεται. 572 υπέρ κατά εγκρίνεται. 573 υπέρ κατά εκπι, ε, απορρίπτεται. 574 υπέρ κατά απορρίπτεται. 575 υπέρ κατά εγκρίνεται. 576 εκπίπτει, 577 Υπέρ. Κατά. Απολύπτεται. 578. Υπέρ. Κατά. 578. 578. Υπέρ. Κατά. Έγκριντ. 579. Κατά. Έλεγχος. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 580. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 8 εκπίπτει. 9 υπέρ Κατά. Έλεγχος. Ναι, ναι. στις προφορίες. Εγκρίνεται. Δέκα Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Κατά εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 28 και 29 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 31 υπέρ κατά εγκρίνεται 32 κατά εγκρίνεται συμβαστική 2 κατά εγκρίνεται 36 υπέρ κατά δεν, είναι εγκρίνεται έλεγχος για 36 Έλεγχος για 36 έρχεται. Πέρας. Σαφές. 42. Κατά. Παρακαλώ. Συγκεντρωθείτε. 42 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 43. Κατά. Εγκρίνεται. 44. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Κατά. Εγκρίνεται. 15 εγκρίνεται. Συμβαστική 4 εγκρίνεται. 62 κατά εγκρίνεται. 63 κατά εγκρίνεται. 64 κατά εγκρίνεται. 65 εκπίτη. Έλεγχος για την 64 πρώτα. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 65. Κατά. Έλεγχος στην 65. Πέρας. Απορρίπτεται 66. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά εγκρίνεται 68 υπέρ κατά εγκρίνεται 69 υπέρ κατά εγκρίνεται 70, 71, 72 υπέρ κατά εγκρίνεται 73 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 6 κατά εγκρίνεται 90 κατά εγκρίνεται 91 κατά έλεγχο στην 91 πέρας απορρίπτεται 92 υπέρ κατά εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 93 και πάλι. Υπέρ. Κατά. Έλεγχο στην 93. Πέρας. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 109. Κατά. Εγκρίνεται. Ρέγγι 27. Την ψηφίσουμε ή όχι. Ρέγγε 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ρέγγε 27 κατά εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά εγκρίνεται. 31 κατά εγκρίνεται. NV1 κατά εγκρίνεται. NV5 κατά απορρίπτεται. NV6 κατά απορρίπτεται. NV9 κατά εγκρίνεται. NV13 κατά εγκρίνεται. Η τελική ψηφοφορία Άρχεται. Πε, πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Επόμενο. Δεν έχουμε καιρό για να κάνουμε πάρτι εδώ πέρα. Τη κυρία Τσαβέλα. Τροπολογία 24. 24. Κατά. Εγκρίνεται. 30. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, μια στιγμή, μια στιγμή, λάθος. Ρέγγια 16. Κατά. Εγκρίνεται. Ρέγγε 20. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Κατά εγκρίνεται. 43. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Κατά εγκρίνεται. 53. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Κατά εγκρίνεται. Κουλτούρα 12. Κατά. Απορρίπτεται. 58 και 59. Κατά. Απορρίπτονται. Συμβαστική 5. Κατά. Εγκρίνεται. Ήμκο 9. Κατά. Εγκρίνεται. Ήμκο 22. Κατά. Εγκρίνεται. Κάλτσο 15. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Κατά εγκρίνεται. Ήλκο 8. Κατά εγκρίνεται. 72 δέλτα και 73 δέλτα είναι ταυτόσιμες κατά απορρίπτονται 75 75 Κατά. Εγκρίνεται. 76. Κατά. Εγκρίνεται. Κουλτούρα 9. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Κατά εγκρίνεται. 88. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Συμβαστική 13. Κατά εγκρίνεται. 97. Κατά εγκρίνεται. 98. Κατά εγκρίνεται. 99 κατά εγκρίνεται. 100 κατά εγκρίνεται. 101 κατά απορρίπτεται. 102 κατά δεκτή. Συμβαστική 14 κατά δεκτή. Ρέκι 21 κατά εγκρίνεται. 105 κατά εγκρίνεται 106 σε δύο τμήματα όχι όχι 106 όλοι μαζί κατά εγκρίνεται 107 κατά εγκρίνεται συμβαστική 15 κατά εγκρίνεται συμβαστική 16 κατά εγκρίνεται Συμβαστική 17. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ρέγγι 19. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Κατά εγκρίνεται. Κατόν

Πέρας. Απορρίπτεται. 121. Κατά. Από εγκρίνεται. 122, 123, 124. Κατά. Εγκρίνονται. 126. Κατά. Απορρίπτονται. 127. Κατά. Απορρίπτονται. Συμβαστική 18 κατά απορρίπτεται. Εγκρίνεται δηλαδή. Έλεγχος, έλεγχος. Έλεγχος για τη 18 συμβαστική. Δεκαοκτώ συμβαστική. Πέρασε. έκπληξη. Μια μικρή έκπληξη. Το έχουμε παρακάνει με τις ψηφοφορίες. 1.32. Κατά. Απορρίπτεται. 1.34. Απορρίπτεται. 1.35 δέλτα κατά απορρίπτεται. 1.36 κατά δεκτή. 1.37 και 38 κατά απορρίπτεται. 1.39 κατά εγκρίνεται. 1.41 κατά εγκρίνεται. 1.43 κατά εγκρίνεται.

κατά. Απορρίπτεται. Ένα πενήντα δύο. Κατά. Δεκτή. Ένα πενήντα. Κατά. Εγκρίνεται. Σήμερα στη δεκαετία. Κατά. Κανεί δεν είναι κατά. Εγκρίνεται. 1.56. Κατά. Εγκρίνεται. 157. Κατά. Εγκρίνεται. 159. Κατά. Εγκρίνεται. Ήμικο 17. Κατά. Εγκρίνεται. Ήμικο 20. Κατά. Εγκρίνεται. Κουλτούρα 3. Κατά. Εγκρίνεται. Κουλτούρα 16 κατά εγκρίνεται. Κουλτούρα 18 κατά εγκρίνεται. Ήμκο 10 κατά εγκρίνεται. 162 κατά εγκρίνεται. 163 κατά εγκρίνεται. 164 κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 κατά εγκρίνεται. 168 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 21 κατά εγκρίνεται. 1,72 κατά απορρίπτεται. 1,73 1,72 απερίφθη. Έλεγχος, 172.

απόλυτο 195 κατά απόλυτο 176 κατά εγκρίνεται ΙΜΚΟ 6 κατά εγκρίνεται 177 κατά εγκρίνεται 178 κατά εγκρίνεται 179 κατά εγκρίνεται τροπολογία 9 κατά δεκτή. Συμβαστική 22 κατά εγκρίνεται. 12 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 23 κατά εγκρίνεται. 24 συμβαστική κατά εγκρίνεται. 19 δέλτα κατά απορρίπτεται. 22 δέλτα είναι ταυτόσιμη, 21 κατά εγκρίνεται. 22 κατά εγκρίνεται. Ρέγγι α κατά εγκρίνεται. Ρέγγι β κατά εγκρίνεται. 1 κατά εγκρίνεται. 2 κατά εγκρίνεται. 4 κατά εγκρίνεται. 5 κατά εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρόνια άρχιτη ψηφοφορία. Κουράστηκε και το μηχάνημα εδώ πέρα. Πέρας. Έχουμε άλλε δύο. Ο Αλάχ, λέει πρόεδρος. Μπράβο, μπράβο. Ομοφωνία. Συγχαρητήρια. Θαυμάσιο αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στην έκθεση Κάλφιν. Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού τι προσωπολογίε υπέρ, κατά, απερίφθησαν 15, υπέρ, απορρίπτεται 16, 16, κατά, εγκρίνεται 2, κατά, εγκρίνεται 17 κατά εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. 5 πρέπει να συνεχίσουμε. Κατά εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά εγκρίνεται. 19 κατά εγκρίνεται. 20 κατά απορρίπτεται. 21 την 20 θέλετε πάλι. Έλεγχος. Έλεγχος για την 20. Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Κατά. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 25 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 26 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 27 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 28 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 29 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 30 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 31 υπέρ. Κατά εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 35 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 37 ε, υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Θέλετε ελέγχο. Εντάξει, για τις 40. 40. Πέρας. Εγκρίνεται 41 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται η 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 6. Κατά. Εγκρίνεται 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 10 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 11. Δεν έχουμε 11 πλάκα έκανα. Τελική ψηφοφορία. Συγγνώμη, ε, συγγνώμη, παστιεύομαι, αλλά τόση ώρα μετά. Πέρας. Καταπληκτικό. Και τώρα τελευταία ψηφοφορία, Beauty είναι σημαντικό. Ένα. Κατά. Ξανά. Ε, έλεγχος ε, για την πρώτη τροπολογία. Απορρίπτεται. 2 κατά εγκρίνεται η συμβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται η συμβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται η 6 κατά εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται και τώρα συμβαστική 5 υπέρ όχι η 5 Συμβαστική 4. 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13. Κατά. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Είναι τμηματική ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 23 υπέρ. 23, αυτό είπα. Ε, κατά. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Ε, έλεγχος για το 26. Ή ε, μάλλον, 26 υπέρ. Κατά έλεγχος. Για το πρώτο τμήμα της 26. Πέρας. Κρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Κατά. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Γκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Ε, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. 30 το 30. Κατά. Εγκρίνεται. Έλεγχος. 30. Έλεγχος για την 30. Δεν αντέχει, τα έχει φτύσει το μηχάνημα. Man and um, adopted. 31. Α, σημαστική 7, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 37 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Έχει κατά. Εγκρίνεται. Και η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Äh, die restlichen Punkte, was machen wir damit? setzen ab